Ωραία που είμαστε όλοι εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή μου ως της, ε, ο πρόεδρος της Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να προεδρεύω σε αυτό το εργαστήριο. Καλησπέρα σας. Είναι χαρά και τιμή μου να προεδρεύω στο πάνελ αυτό ε, υψηλού επίπεδου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Σας ομιλώ από τις ε, Κανάριες ε, νήσους όπου η κατάσταση εδώ παρέχει ίσως κορυφωθεί στην πιο επικίνδυνη διαδρομή αυτή του Ατλαντικού ωκεανού. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να εκμεταλλευτούμε αυτήν την συζήτηση. Με χαρά μου καλωσορίζω την Επίτροπο Ιστορικών, την κυρία Γιωχάνσεν και τον κύριο Χώσε Χόφερ, Υπουργό Ιστορικών της Γερμανίας που εκπροσωπεί την Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά θα ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Χρήστο, ε, Διεθνή Πρόεδρο των Ιατρών Χωρίς ε, Σύνορα που θα μας μιλήσει για την ανθρωπιστική διάσταση. Το θέμα το οποίο συζητάμε σχετίζεται με την εντολή που υπάρχει στην συνθήκη της Λισαβόνας του άρθρο 80 περί αλληλεγγύης και κοινή ευθύνη και στην ε, χάραξη της πολιτικής ε, και στην ε, νομοθεσία για ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Η αρχή της αλληλεγγύης ε, και της ε, κοινή ευθύνη δεν είναι μόνο υποχρέωση της ε, συνθήκης, αλλά και πυλώνας του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου. Όμως έχουμε συναντήσει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες στην προσπάθειά μας να καταστεί το πραγματικό. Θα ακούσουμε τώρα την μαρτυρία από δύο σημεία που είναι στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης από τους δημάρχους ε, και Λαμπεντούζας. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να δούμε μια μαρτυρία για μια εμπειρία η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό, εδώ και πέντε χρόνια. Δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ, θα μας τα πούν, είμαι σίγουρος. Εγώ θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε την λεγόμενη ολιστική προσέγγιση για άσυλο και μετανάστευση. Ε, δηλαδή για αλληλεγγύη αλλά και για δράσεις στις χώρες προέλευσης ε, και διέλευσης και στις χώρες προορισμού βεβαίως της μετανάστευσης ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης και των ευκαιριών αλλά βεβαίως ε, χωρίζοντας ε, κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ ε, της ε, παρατυπής μετανάστευσης και όσων δικαιούνται άσυλο οπότε η προσέγγιση αυτή πρέπει να μιλήσει και για επιστροφές Ελπίζω λοιπόν να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και μια ευκαιρία να δούμε τις προσδοκίες που προκύπτουν από το νέο σύμφωνο το οποίο έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Ελευθεριών από την Επιτροπή την κυρία Γιωχάνσεν την οποία θα ακούσουμε επίσης και ακούσουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου για το τι κάνει ο κύριος Ζέχοφερ. Για είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, είναι πολύ πρακτική. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε οι αρχές ε, και οι αξίες ε, που αναφέρονται στο χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύουν ε, όσους βρίσκονται στο ευρωπαϊκό έδαφος παρά το ότι μπορεί να μην είναι ευρωπαίοι πολίτες γιατί είναι άνθρωποι είναι κάτι το ουσιώδες. Και εκφράζουμε την ανησυχία της Επιτροπής μας για το κράτος και είμαι σίγουρος ότι ο δόκτωρας Χριστός Χριστού θα μας διαφωτίσει για αυτά. Πριν όμως δώσω τον λόγο, καλωσορίζω τον Ανδρέα Λίνχοτς, πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής της ε, Γερμανικής ε, Βουλής. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Κυρία Λιντχόλτς. Αξιότιμη κύριε Αγγιλάρα, αξιότιμη κύριε Επίτροπε Γιώχανσεν, κύριε Ζέχοφερ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά από το Βερολίνο να σας απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσατε να έρθετε κι εσείς σε αυτήν την συνάντηση. Το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις γενικές πτυχές ε, μιας κοινή ε, πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο και το πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε δούμε αυτή την πολιτική. Το ε, επόμενο αυτό διάστημα της μια μισή ώρα θα δούμε τα θέματα της αλληλεγγύης ε, και της ευθύνης ό,τι αφορά την διαχείριση της ε, κρίσης. Αλληλεγγύη είναι ο συνδετικό ιστό ουσιαστικά που θα πρέπει τουλάχιστον να συγκρατεί μεταξύ του τα κράτη-μέλη. Από τι 9 Μαου του 50 με τη δήλωση Σουμάν, η αλληλεγγύη είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η Ευρώπη ε, δεν πρόκειται ε, να ε, γίνει από μόνη της αλλά με συγκεκριμένα επιτεύγματα και το βασικό είναι να γίνει αυτό μέσω αλληλεγγύης, αλληλεγγύη λοιπόν. Και είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα υπάρχει πραγματικά στις πράξεις, στα έργα αλληλεγγύη, γιατί αυτό ζητούσε ο Σουμάνι το 50 έμπρακτα αλληλεγγύη και Έχουμε πολύ δύσκολα ζητήματα να λύσουμε τη μετανάστευση στο άσυλο. Πρέπει να βρούμε λύσει ε, και είμαστε κάπω μετέωροι όλο αυτό το διάστημα των τεσσάρων χρόνων. Τα τελευταία χρόνια μα έδειξαν ότι αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ε, αλληλεγγύη υποχρεωτική δεν θα προχωρήσουμε. Είδαμε επίση ότι δεν είναι δυνατόν κάθε ευρωπαϊκό κράτος ε, φυσικά να έχει την ίδια ακριβώς συμμετοχή. Χρειάζεται ένα ευέλικτο σύστημα αλληλεγγύης ε, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει δώσει αυτή τη βάση συζήτηση. Ε, στα κράτη-μέλη γίνεται πολύ σημαντική συζήτηση. Είναι διαφορετικός ο φόρτος, διαφορετική γεωγραφική θέση της κάθε χώρας και τη μορφολογία της. Υπάρχουν μετανάστες που έρχονται στην Ένωση από συγκεκριμένε χώρες. Υπάρχει επομένως ε, η ανάγκη να υπάρξει ε, επιμερισμός των βάρων και επίσης ε, με τη συνοριαφυλακή, φυλακή, με οικονομικούς πόρους μπορούμε να συνδράμουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι καλό το ότι έχουμε τώρα μια επιταχυμένη, βούλησε τουλάχιστον μια επιταχυμένη πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο και να έχουμε και βέβαια το θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, ε, ε, την κλίδα ε, στη, στα εσωτερικά σύνορα. Θέλουμε επίσης οι διαδικασίες να είναι σύμφωνα με το κράτος δικαίου, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Έχουν κάνει πολύ καλές προτάσεις υπηρεσίες κομισιών και θα πρέπει να δούμε τώρα με τις ασύλου πώς όλα αυτά θα τα διεκπαιρεώσουν. Υπάρχουν καλές προτάσεις. Στην πράξη όμως είναι το θέμα πώς θα εφαρμοστούν γιατί η έμπρακτη εφαρμογή είναι το δύσκολο δύσκολο όπως είδαμε πολλές φορές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να λογοδοτήσουμε, ε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ε, δραστηριοποιούμαστε για τη μετανάστευση, αλλά δεν πρέπει να δοθούν και λάθος κίνητρα σε κάποια κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σομερής επιμερισμός των βαρών. Θεωρούμε τέλος σημαντικό να ε, τελειώσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου ε, σύντομα και ε, πιστεύω ότι συμφωνεί και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση ε, μόνο όταν υπάρχει συνοχή ε, και ενότητα στα κράτη-μέλη για να έχουμε την ολοκλήρωση, την ένταξη. Θα ευχαριστήσω όλους τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν βάλει και αυτό λιθαράκι τους για την ένταξη των ατόμων οι οποίοι έρχονται στις χώρες μέλη της Ένωσης. Και ένα τελευταίο σημείο εισαγωγικά που φαντάζομαι ότι θα εμβαθύνεται στην συζήτηση που θα ακολουθήσει και ε, αφού ακούσουμε βέβαια και τους, ε, τον κύριο Ζεχόφερ, την κυρία Γιώχανσον ε, θα έρθουμε σε ένα γύρο έρωτα απαντήσεων. ένα μισή λεπτό θα είναι ο χρόνος που θα δίνουμε για την κάθε ερώτηση γιατί είναι πολλές ερωτήσεις. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω και γι' αυτό μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Δεν το λόγο στην κυρία Γιώχανσον, την Επιτρόπο. Thank you. Thank you very Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την μετανάστευση. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Η μετανάστευση είναι μια κανονικότητα. Η μετανάστευση πάντοτε υπήρχε, θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν είναι κάτι πολύ να φοβόμαστε. Η μετανάστευση είναι κάτι που πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι κάθε χρόνο Έχουμε πολλούς νόμιμους μετανάστες προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι, 3 εκατομμύρια μετανάστες ήρθαν εδώ νομίμως. Οι περισσότεροι, διότι ε, είχαν κάποια σχέση με, και ερωτεύτηκαν Ευρωπαίο πολίτη για άλλους οικογενειακούς λόγους. Ήρθαν για να εργαστούν πάνω από ένα εκατομμύριο πέρσι, έρχονται για να σπουδάσουν, για έρευνα ε, ή κάποιοι επειδή διεθνού διεθνούς προστασία. Κάθε χρόνο ένα-ενάμιση εκατομμύριο κόσμο αφήνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω του. Κυρίω γιατί και πάλι δοτεύτηκαν ε, κάποιον εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ή για άλλου οικογενειακού λόγου ή για να δουλέψουν. Ε, υπάρχει ένα πηγενέλα κάθε χρονιά και αυτό είναι καλό γιατί χρειαζόμαστε μετανάστε και είμαστε μια γυράσκουσα κοινωνία. Οι περισσότεροι που έρχονται μπορεί να μείνουν ε, για πάντα σχεδόν. Πέρσι μόνο 700.000 πήραν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και αυτό είναι είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι είναι τεράστιο κομμάτι του φαινομένου τη μετανάστευση αυτό. Υπάρχει ένα άλλο μικρότερο τμήμα ανθρώπων που έρχονται ατύπω. Πέρσι είχαμε 140.000 ε, παράτυπου μετανάστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση για τη μετανάστευση έχει δυστυχώς πέσει θύμα εδώ και πολλά χρόνια ε, μιας ε, τραγώδησης ε, του τι συμβαίνει. Θα πρέπει να βγει αυτός ο δραματικός τόνος από την όλη συζήτηση τη μετανάστευσης αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα ψύχρεμα. Ε, η κατάσταση για τους μετανάστες μπορεί να είναι όντως δραματική. Ε, σε κάποια ευρωπαϊκά νησιά επίσης η κατάσταση είναι δραματική. Πρέπει να το πούμε. Ωστόσο η συζήτηση περί πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθεί ε, σε θέματα άνευ δραματικού τόνου και να είμαστε διαυγείς και αντικειμενικοί αν θέλουμε να βρούμε λύσεις. Το πιο σημαντικό πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε να προασπιστούμε και να προστατεύσουμε το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου. Είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι μέρος των αξιών μας, ε, γράφεται και στις συνθήκες μας και στις συμβάσεις ε, στις οποίες έχουμε συμπληθεί. Άρα είναι η βάση για τις προτάσεις που θα συμπεριληφθούν στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή πρέπει να, εργαζόμαστε πολύ, ε, να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τρίτες χώρες. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με τις χώρες εταίρους μας για να τις ενισχύσουμε. Εκείνες που υποδέχονται πολλούς πρόσφυγες λόγω χάρη σήμερα πρέπει να τους δείξουμε αλληλεγγύη, πρέπει να εργαστούμε και να συνεργαστούμε στενά με ε, χώρες για να αντιμετωπίσουμε τους εμπόρους και τους λαθρεμπόρους ανθρώπων, να βεβαιωθούμε ότι παίρνουν πίσω τους δικούς τους πολίτες αφού πρέπει να επιστραφούν και να τους βοηθήσουμε να κάνουν στρατηγικές επενδύσεις και να χτίσουμε μέσω του μετανάστευση. Η εξωτερική διάσταση λοιπόν είναι τεράστιο θέμα για τη μετανάστευση. Αλλά ήθελα εδώ να επικεντρωθώ στις ελλείψεις του ευρωπαϊκού συστήματο, αυτέ που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με το νέο σύμφωνο. Τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα οι παράνομε αφήξει. Δεύτερον οι επιστροφέ και τρίτον η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις παράνομες αφήξει. Ε, Όπω είπα πέρσι, είχαμε 140.000 παράτυπε αφήξει. Οι περισσότερε από αυτέ ε, ήταν αφήξει ανθρώπων που έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του για να έρθουν ω εδώ και πλήρωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσό σε οργανωμένα δίκτυα, ισχυρά και πολύ καλά διαρθρωμένα ε, παράνομα δίκτυα για να φτάσουν λαθρέως εδώ. Πρέπει να μειώσουμε τις ε, παράνομες αφήξεις και ανταυτού να έχουμε περισσότερες νόμιμες αφήξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε λιγότερου μετανάστε. Χρειαζόμαστε όμω περισσότερου νομίμου μετανάστε. Να έρχονται από τι νόμιμε οδού. Και πρόσφυγε ενδεχομένω και αυτού που θέλουν να συμβάλλουν και στην οικονομία μα. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στην επικατάσταση. Γι' αυτό κοιτάζουμε και ένα πρόγραμμα μετεγκατάσταση ε, που θα το ε, στηρίζει η κοινότητα, η Ένωση. Και θα δημιουργήσουμε τι κατάλληλε νόμιμε οδού. Αλλά πρέπει να καταπολεμήσουμε και του λαθρεμπόρου. Ε, κάτι που πρέπει να το κάνουμε σε συνεργασία με τι χώρε εταίρου, τι τρίτε χώρε. Ε, δεύτερον, οι επιστροφέ. Όταν ε, μιλώ στου Ευρωπαίου πολίτε, συνειδητοποιώ ότι οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν αυτούς που χρήζουν ε, διεθνού προστασία και είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν αυτού που θέλουν να συμβάλλουν θετικά στην οικονομία μα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ όσων είναι ε, επιλέξιμοι για να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είναι θερμό το καλό όρισμά μα προ αυτού και θα πρέπει να του επιτρόψουμε την ένταξή του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία. Αυτοί όμω που δεν είναι επιλέξιμοι και δεν μπορούν να παραμείνουν πρέπει να επιστραφούν. Σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία όσων έρχονται παρανόμως δεν χρήζουν διεθνούς προστασίες. Θα πάρουν αρνητική απόφαση στην αίτηση ασύλου τους και θα πρέπει να ε, επιστραφούν. Πρέπει λοιπόν εδώ να μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα σύστημα. Ένα σύστημα για να μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν. Αυτός ε, είναι και ο λόγος που θέλουμε να έχουμε νόμιμες οδούς. Θα πρέπει να ε, φεύγουν αυτοί που ε, παρανόμως βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, αν δεν επιστραφούν εμποδίζονται και νόμιμοι οδοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο τρίτων χωρών. Ε, σε αυτό έχω επικεντρωθεί αυτόν τον καιρό. Και μετά είναι και η ελληνική μεταξύ των κρατών μελών ως τρίτο. Είναι σαφές ότι οι παράνομες αφήξει σε κάποιες χώρες ε, είναι πολύ περισσότερες από τις άλλες. Είναι ε, ουσιώδε να δείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ των 100 μελών εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή μου, η, η οικειοθελή επίδειξη αλληλεγγύη δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχουν να υπήρξε ένα ε, δεσμευτικό μηχανισμό αλληλεγγύη και αυτό έχουμε προτείνει στο σύμφωνό μα. Είναι βέβαια ότι μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη με διαφορετικού τρόπου, λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση του τι συμβαίνει. Ε, εάν οι πλειοψηφίε σου φτάνουν πρέπει να επιστραφούν. Επίση, μπορεί να υπάρξει μια ιδέα ε, συνδρομή μεταξύ κρατών μελών για την επιστροφή κάποιων ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μπορέσουν κάποιε χώρε να επιστρέψουν στι χώρε καταγωγή του κάποιου ανθρώπου πραγματικά. Και μετά είναι και με την κατάσταση αυτό. Είναι σημαντικό για να ε, μπορέσουν να επιστραφούν σωστά όσοι ε, χρήζουν διεθνούς προστασία ή όχι. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ταχύτερη διαδικασία γιατί ε, το καθοριστικό στοιχείο εδώ είναι ο χρόνος. Εάν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στις επιστροφές μας και την επανένταξη που είναι και αυτό σημαντικό μέρος των επιστροφών. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι το σύμφωνο που έχουμε προτείνει είναι μια συμβαστική λύση βεβαίω, είναι μια εξισορροπημένη λύση. Διότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικέ πραγματικότητε. Κάποιε είναι χώρε πρώτη άφηξη, κάποιε είναι χώρε προορισμού ε, δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι πολύ διαφορετικέ οι γεωγραφικέ του συνθήκε. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να λάβουμε διαφορετικά μέτρα ανάλογα με το κράτο μέλο. Επίση, υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει και για άλλου λόγου ότι αφορά τη μετανάστευση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι ε, εμεί ε, οι πολιτικοί μπορούμε να κάνουμε τι απαραίτητου συμβιβασμού ε, για να βρούμε λύσει, να βγούμε από τα διέξοδα και να προβλέψουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα αλληλεγγύη και ευθύνη ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι να πω ότι δεν είναι ε, δυνατό για όποιον το επιθυμεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, έρθει και να μείνει. Ούτε όποιο θέλει να μπει μπορεί και να παραμείνει. Όμω όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι μετανάστε είναι ε, άνθρωποι, είναι ανθρώπινα όντα. Παρόλο λοιπόν που πρέπει να επιστραφούν ενδεχομένω κάποιοι άνθρωποι, παραμένουν ανθρώπινα όντα. Έχουν δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, ε, τους μεταχειριζόμαστε βάσει των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπεια τους, ασχέτως του αν έχουν πραγματικά δικαίωμα να παραμείνουν ή όχι. Ευχαριστώ. Äh, σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιώχανσεν για την εισαγωγή σας αυτή η παρέμβαση και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ζέχοφερ, καθότι η Γερμανική Προεδρία προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο σε αυτή την ε, κοινή προσπάθεια μετανάστευση. Περιμένουμε εναγωνίω την παρέμβασή σα. ich vielleicht vorschlagen, dass wir... Να ήθελα να προτείνω να περάσουμε αμέσως στον δόκτωρα Χρήστο Χρήστο πρόεδρο των γιατρών χωρίς σύνορα μας ακούτε Α,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 Äh, er- Θα επιστρέψουμε στον Υπουργό των Ιστορικών. Δεν έχουμε σύνδεση αυτή τη στιγμή μαζί του. So, Sie müssten mir jetzt sagen, mit wem wir es probieren könnten. Entweder... Λοιπόν, με ποιον μπορούμε. Με τον Υπουργό ή με τον κύριο Χρήστο. Ας δοκιμάσουμε με τον κύριο Ζέχοφερ. Herr Seehofer? Sie können jetzt sprechen. Μιλήστε. Δυστυχώς δεν έχουμε ήχο. The next speaker, Mr. Christo, would be a... Ο κύριος Χρήστο είναι διαθέσιμος. Okay, I take over then. And uh, thank you very much. It's really a Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να δώσουμε και εμείς την δική μας την άποψη, η οποία διαμορφώθηκε από την εμπειρία αυτών που πεθαίνουν προσπαθώντας να φτάσουν σε κάποια ασφαλεία. Ε, έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι στην ε, Μεσογείο μεταξύ των οποίων και ένα μωρό τελευταία και το πλήρωμα του πλοίου Open Arms της μόνης ΜΚΟ που δρά ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Στην Ελλάδα ένας πατέρας έχασε το εξάχρονο παιδί του και τελικά συνελήφθη επειδή το εξέθεσε σε κίνδυνο και αντιμετωπίζει φυλάκιση 10 ετών. Ε, δηλαδή δεν έχει υποφέρει αρκετά. Εφτά νεαροί Βόρειο Αφρικανοί βρέθηκαν σε ένα κοντέινερ στην Παραγουάη. Προσπαθούσαν να πάνε στην Κροατία, αλλά μετά από διάφορες αποθήσεις αποφάσισαν να μπουν σε ένα κοντέινερ, νομίζω ότι θα φτάσουν στο Μιλάνο. Ε, τα πτώματα τα βρήκαν ε, σε αποσύνθεση μετά από τέσσερις ε, μήνες. Πέθαναν από την πείνα. Οι θάνατοι αυτοί όπως και η φρίκη των ελληνικών ε, εγκαταστάσεων δεν είναι κάποιο ατύχημα ανεξήγητο είναι άμεση συνέπεια πολιτικών όπως ε, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η παρέτηση από την ε, ευθύνη για διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης σε διεθνή ύδατα και σε ευρωπαϊκά ύδατα. Ε, δηλαδή πρέπει να τα δεχτούμε αυτά έτσι ως κάποιες ε, συνέπειες. Ε. Εγώ θεωρώ όχι. Αυτό το οποίο λοιπόν ζει η Ευρώπη δεν είναι μια ανθρωπιστική κρίση, είναι μια κρίση ανθρωπισμού. Η σημερινή συνεδρίαση μιλάει για αλληλεγγύη, αλλά πού βρίσκεται η πραγματική αλληλεγγύη. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη κάνουν κατάχρηση του όρου. Έχουν αποτύχει στη συλλογική του ευθύνη να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή έχουν χρησιμοποιήσει και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ κρατών για να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Αλληλεγγύη δεν σημαίνει παζάρι μεταξύ κρατών για το ποιος θα πάρει πόσους, με ποια τιμή κτλ. Μια προσπάθεια να βρεθεί πολιτικός συμβασμός έχουν παραμεληθεί οι ανάγκες ανθρώπων. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι ομάδες μας ε, εργάζονται άοκνα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πιο οδυνηρές συνέπειες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές οι οποίες είναι άμεσα υπεύθυνε για αυτήν την φρίκη. Ξανά και ξανά δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θεώρησαν αυτό ευκαιρία για να σταματήσουν να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε άρνηση οι επίσημες δηλώσεις ε, περί τραγωδιών ε, βαλκανικής ε, διόδου ή της φρίκης των στρατοπέδων κράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ότι αυτά έχουν γίνει με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μετά από τις φωτιές στη Μόρια ακούσαμε όχι άλλη Μόρια. Τι σημαίνει αυτό όμως όταν βλέπουμε τέτοια στρατόπεδα σε όλα τα νησιά, στη Σάμο, στη Λέσβο, στην στη Χίο, στη Λέρο χρόνο με το χρόνο μας λένε ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες αλλά συνέχεια το προσωπικό μας βλέπει την ε, επιδίνωση της υγείας ε, των ανθρώπων αυτών που κοιμούνται κάτω από τις ελιές. Και ενώ χαιρόμαστε για την περιορισμένη ανακατανομή κάποιων ανηλίκων και ασυνόδευτων ανηλίκων οι προσπάθειες αυτές είναι ένα μικρό τμήμα της λύσης. Πώς μπορούν να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές εκατοντάδες άτομα την ίδια στιγμή που αναπτύσσει ένα σύστημα αποτροπής που θα έχει τις ίδιες συνέπειες. Η νέα αυτή απάνθρωπη κανονικότητα έχει γίνει αποδεκτή και στην κεντρική Μεσόγειο. Εδώ οι ηγέτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοούν τις διεθνείς υποχρεώσει τους για έρευνα και διάσωση. Δεν χρησιμοποιούν ε, ευρωπαϊκά σκάφη κοντά στις ακτές ε, και εύκολα συμφώνησαν ε, με το να αφήσουν την έρευνα και διάσωση στην Λιβική ακτοφυλακή. Ως αποτέλεσμα αυτού, 100.000 άτομα έχουν αναχαιριστεί και επιστραφεί στην Λιβύη τα τελευταία χρόνια και εκεί πέρα αντιμετωπίζουν ε, απάνθρωπες συνθήκες, ε, κρατήσεις, ε, εκμετάλλευση. Οι αρχές της Λιβύης έχουν πραγματικά καταστροφικό ιστορικό στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος φαίνεται ότι είναι ότι θέλουν να τους αποτρέψουν να έρθουν στις Ευρωπαϊκές Ακτές με οποιοδήποτε κόστος όμως οι δράσει της Ευρωπαϊκή Ένωση εκτείνονται και πέρα από τα σύνορά τη. Έχουμε μια εκστρατεία συκοφάντησης και παρεμπόδισης ε, των ΜΚΟ. Οι γιατροί χωρίς σύνορα και άλλοι έχουν ε, υποστεί αστήρικτες κατηγορίες, ε, μας λένε διακινητές, ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τεχνικές προδιαγραφές. Πρόκειται για μια ενορχιστρωμένη εκστρατεία που έχει πραγματικά αποδεκατήσει τις προσπάθειες ε, πολιτών. Αυτή τη στιγμή έξι πλοία έχουν δεσμευτεί σε Ιταλικά λιμάνια και συνεχώς εφευρίσκουν νέους λόγους για να μην τα αφήσουν να αποπλέψουν. Η Κομισιόν ε, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό οι προστασίες του νέου συμφώνου είναι πολύ ασθενείς και επιπλέον νομοποιούνται οι φυστάμενες πρακτικές που έχουν γίνει αντικείμενο κατάχρησης για να σταματήσει η παρουσία των ΜΚΟ. Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλουν να σώσουν σώες στην θάλασσα, τουλάχιστον να, να μην σταματάνε τις ΜΚΟ. Συμπερασματικά. Αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή και αν η Ευρώπη δεν αναλάβει τις ευθύνες της, θα έχουμε... Κύριε Χρήστο, πρέπει να τελειώνετε. Έχετε μιλήσει ήδη δύο φορές περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί. Mr. you can press the click. Uh Κύριε Ζεχόφερ, πιέσατε το κονδύον. Äh, τρίτη προσπάθεια, τρίτη και καλή. Δυστυχώς πάρα πολύ χαμηλά ο ήχος. Κύριε Ζεχόφερ, ε, συγγνώμη σας διακόπτω λέει συντονίστρια, αλλά είναι πολύ χαμηλός ο ήχος σας, δεν ακούγεστε αρκετά. Way to increase your volume. Die Lautstärke ist leider Μπορείτε να βάσετε λίγο τον ήχο του μικροφόνου σας. Είναι καλύτερα τώρα. Ja, wir können das so versuchen. Προσπαθήσουμε έτσι. Τέταρτη προσπάθεια. Θα με καταλαβαίνετε. Αν μιλάμε ψιθυριστά μπορεί να ακούμε οι διερμηνείς. Αγαπητή Αντρέα, αγαπητέ Πρόεδρε Χουάν Φερνάντο, αγαπητή Επίτροπε Ήλβα, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι αλήθειες θα ήθελα να πω στην αρχή της παρέμβασής μου. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι η μετανάστευση για πολλά πολλά ακόμη χρόνια θα μας απασχολεί στην Ευρώπη. Δεύτερη αλήθεια, τα μεταναστευτικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την μελλοντική ικανότητα και δυνατότητα και της Ένωσης. Και το τρίτο, τρίτη αλήθεια, Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ε, βρει μια βιώσιμη απάντηση στην αντιμετώπιση του ζητήματος και αν δεν βρούμε τότε η κλιμάκωση θα ε, συνεχίσει ε, και θα ωφελήσει αυτούς που είναι αντίθετοι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτά είναι τα στήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μία δέσμη μέτρων συζήτηση και η Επίτροπος σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύση που θα είναι 100% ε, ικανοποιητική για όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τα κράτη που έχουν τα εξωτερικά σύνορα, ε, που είναι οι χώρε πρώτη άφηξη, και αυτοί μα ζητούν περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πρέπει να την εξασφαλίσουμε. Υπάρχουν τα κράτη Βίζεγκρατ ε, και άλλα που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με την έννοια της αλληλεγγύης και απ' την άλλη έχουμε τις χώρες στο κέντρο της Ευρώπης ε, που πολύ σωστά περιμένουν ότι δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις στο σύστημα της ε, μετανάστευσης και του ασύλου. Η δική μου προσωπική πεποίθηση και είναι η δεύτερη δεκαετία που ασχολούμαι με το θέμα αυτό στην πράξη θεωρώ ότι το κλειδί θα είναι μια πιο αναλογική σχέση μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, τα κράτη της Νότιας Ευρώπης αν τα απαλλάξουμε αισθητά από το βάρος τους ε, και έτσι ε, θα μπορέσουμε να έχουμε αυτήν την δόση ε, ευθύνης από την πλευρά τους και αλληλεγγύης από την πλευρά μας. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τους νομίμους του άσυλο, αλλά είναι δύσκολη η εξίσωση που έχουμε να λύσουμε για να βρούμε ισορροπίες Πρέπει δηλαδή να έχουν αποτελεσματικές διαδικασίες ε, στα εξωτερικά σύνορα και υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ιδίω ε, αυτές που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το είδαμε προσφάτως ε, και πολλές φορές μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν με τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και στη φωτιά, στην πυρκαγιά, στον καταβλισμό της Λέσβου. Θεωρώ ότι είναι και τα δύο λοιπόν και οι δύο πτυχές σημαντικές, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε ε, τη σωστή προστασία ε, και να την εξασφαλίσουμε σωστή προστασία ε, πρέπει να υπάρχει προστασία στα εξωτερικά σύνορα, να δούμε εκεί πώς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται ε, διεθνούς προστασίας. Εκεί θα πρέπει να γίνει το έλεγχος και έπειτα στη συνέχεια Ευρώπη θα πρέπει συνολικά να δείξει αλληλεγγύη και αυτή να μην περιορίζεται σε λίγα ε, μόνο κράτη τα οποία θα παίρνουν ε, το περισσότερο βάρος. Και γι' αυτό σε ό,τι αφορά την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ε, δηλαδή να έχουμε και μια επαφή με τις χώρες προέλευσης, τις χώρες καταγωγής, να υπάρξει μια συνεργασία. Η Επίτροπος έχει μέχρι στιγμής ε, κάνει ό,τι πρέπει και τα έχει καταφέρει πολύ καλά και Βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε που είναι η πανδημία ε, που χτυπά ε, ακόμα πιο βαριά την Ευρώπη. Και υπάρχει όμως ε, κόσμος που χρειάζεται να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για αυτούς τους λόγους της κρίσης. Όλο αυτό δεν είναι κάτι που αντολίσουμε μόνοι μας. Τρέχει ο χρόνος, κάνουμε μια νέα προσπάθεια επί τη βάση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση ε, είχαμε δύο συμβούλια τα οποία προσπάθησαν και νομίζω ότι πολύ λογικά συζήτησαν ε, το θέμα και νομίζω ότι στόχος μας, στόχος της Γερμανικής ε, Προεδρίας τουλάχιστον και συμφωνούμε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι τουλάχιστον επί της δικής μας Προεδρίας να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική συνεννόηση σε ό,τι αφορά τη βασική αρχιτεκτονική της πολιτικής ασύλου και στην επόμενη Προεδρία να έχουμε την απαραίτητη νομική πράξη. Ε, με τελευταία μέρα της Γερμανικής Προεδρίας, ε, με όλοι μας ε, τις δυνάμεις, θα επεξεργαστώ αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μια ακόμη ημερομηνία, ένα ραντεβού με το Συμβούλιο Εκοφήν, αρχές Δεκεμβρίου προβλέπεται επίσης και πριν από τα Χριστούγεννα στις 13-14 ε, Δεκεμβρίου και ένα άλλο ε, ε, συμβούλιο και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να, να προσυπογράψουν το έγγραφο και 27 χώρες μέλη της Ένωσης. Είμαι αισιόδοξο, παραμένω αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και αυτό θα αποτελέσει ένα τεράστιο μήνυμα. Ένα δείγμα αλληλεγγύης ότι οι Ευρωπαίοι μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που δείχνει αλληλεγγύη και απ' την άλλη κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει τις ευθύνες του, αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Σας ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Χρήστο. Κύριε Υπουργέ Σιχόφερ, ευχαριστώ και τους δυο σας για τις δηλώσεις σας και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Αγγιλάρ. Ε, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους Ευρωβουλευτές που έχουν συνδεθεί, άκουσαν τους ομιλητές μας και θέλουν να πάρουν το λόγο. Ακούσαμε την κυρία Γιώχανσον, τον κύριο Σιχόφερ, τον κύριο Χριστού, ε, πρόεδρο της ε, Medicine Sans Frontières. Εγώ θα ήθελα να θέσω τα εξής θέματα επιτάπητος. Πρώτα απ' όλα τις ελλείψεις του ισχύοντος δικαίου για τη μετανάστευση και το άσυλο, την έλλειψη αλληλεγγύης και την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος, ένας μηχανισμός μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας ή με, ε, με αλλαγές αυτήν ε, για να υπάρξει υποχρεωτική αλληλεγγύη. Πρέπει να δούμε και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση του όλου θέματος. Γιατί από τη μια έχουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε προέλευση, αλλά και τι χώρε διέλευση. Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο τη μετανάστευση. Είναι ένα γεγονό η μετανάστευση. Δεν είναι απειλή, δεν είναι ρίσκο, όπω εξήγησε σωστά η Επιτροπό Γιώχανσον. Και πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε ολιστικά, σφαιρικά ε, μέτρα, με μια πολιτική ακριβώς ολιστική για να έχει νόημα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ε, σωστή και βάση των ευρωπαϊκών κανόνων και νόμων. Και για να είμαστε και συνεπείς, θέλουμε μια πολιτική που να βασίζεται στις, ε, στα δικαιώματα των ανθρώπων, όλη η ευρωπαϊκή εμπειρία, όλο το ευρωπαϊκό εγχειρήμα βασίζεται στο κράτος δικαίου, ε, τα δικαιώματα των ανθρώπων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα παρακαλέσω όλους τους ομιλητές να παραμένουν σε ένα λεπτό ο καθένας, ιδάλλως μπορεί να μην προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπράνκο Σας έχω στον κατάλογο αγορητών μου, κύριε Μπράνκο. Έχετε το λόγο. Κύριε Λόπες Αγγιλάρ, ο κύριος Μπράνκο δεν είναι συνδεδεμένος και η κυρία Εστρέλα δεν είναι και εκείνη. Κύριε Ιτχιτβέγγι, είστε συνδεδεμένος, εάν ναι, σας ακούμε. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ε, το πρωί ακούσαμε μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την κυρία Φοντερ Λάιεν, τον κύριο Σασόλη και άλλους. Ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές τους και την Επίτροπο βεβαίω. Ακούσαμε όμως ε, μία διάσταση να διατρέχει όλες τις παρουσιάσεις περί μετανάστευσης, θεωρώ με έναν τρόπο υπεραπλουστευτικό να παρουσιάζουμε τα πράγματα. Δεν δόθηκε πολύ προσοχή στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και που προκαλεί η μετανάστευση. Δεν ε, αποφεύγουν όλοι οι συνθήκες φτώχειας ή εμπόλεμες σε χώρες με δυσκολίες, στην Αφρική ας πούμε. Κάποιοι έρχονται για οικονομικούς λόγους στην Ευρώπη ξεκάθαρα. Πρέπει να κάνουμε όμως μια σαφή διάκριση μεταξύ των προσφύγων που ε, ζητούν άσυλο και έχουν δικαίωμα στο άσυλο και αυτούς που δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα και θέλουν απλώς να έρθουν ως ε, μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες. Εκεί θα πρέπει να μπορεί να αποφασίσει το κάθε κράτος αν θέλει να τους δεχτεί ή όχι και να έρθουν και αυτό να ε, λαμβάνεται ως απόφαση πρωτού φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τις μεταναστευτικές πολιτικές ως απειλή και ε, κατά της ασφαλείας μας και αυτό έχει προκαλέσει χάος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα του ασύλου έχει γίνει προβληματικό και είδαμε τις επιθέσεις στην Νίκαια, τη Βιέννη και αλλού πρόσφατα ε, ε, και πράχθησαν από μετανάστες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ευθύ. Πρέπει να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα τους Ευρωπαίους πολίτες. Εάν η παράνομη μετανάστευση ε, είναι μια απειλή, δεν θα μπορούμε να τη δεχτούμε. και το θέμα είναι να δούμε ποιοι μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και χρήζουν διεθνούς προστασία. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα δεν θα πέφτει θύμα, δεν θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και δεν θα το χρησιμοποιούν δολίως ε, και θα έρχονται αυτοί που πρέπει να έρθουν. Και το θέμα τη αλληλεγγύη, τελευταία μου παρατήρηση. Πρέπει να είμαστε και εκεί διαλλακτικοί. Διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσει κανεί την αλληλεγγύη του. Η Ουγγαρία έχει εκφράσει την αλληλεγγύη τη προ του Ευρωπαίου εταίρου τη, ε, προστατεύοντα τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Δαπανούμε πολλά κονδύλια. Αυτή είναι η επιπλέον προσπάθειά μα. Αυτή είναι η αλληλεγγύη μα προ την Ευρώπη. Εκεί πρέπει να φανούμε και λίγο διαλλακτικοί. Ε, και για όσους δεν έχουν δικαίωμα στο άσυλο και έρχονται παρόλα αυτά παρανόμως θα πρέπει να επιστρέφονται αμέσως στη χώρα τους. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πρέπει κάποια αρχή να υπάρχει και αυτή είναι η αρχή της λύσης που πρέπει να είναι ρεαλιστική και είναι και απλό να πραγματοποιηθεί. Ε, Α μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει αυτή η κρίση στην Ευρώπη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μετανάστευση που να βασίζεται στην ε, πραγματικότητα, τον πραγματισμό και μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Χιτβέγγι, αλλά για τους υπόλοιπους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου, ε, επειδή είστε πολύ και ο κύριος Χιτβέγγι μίλησε σχεδόν τρία λεπτά, παρακαλώ βιαστείτε λίγο παραπάνω, δεν θα προλάβουμε. Πριν προχωρήσουμε στους υπόλοιπους ε, παρεμβαίνοντες, σας ακούσουμε πρώτα δύο μάρτυρες ο κύριος Στρατής Κιτέλης, ε, δήμαρχος ε, της Μετιλίνης στη Λέσβο και ο κύριος Μαρτέλο, που είναι δήμαρχος της Λαπεντούζα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Κιτέλη, τον δήμαρχο της Μετιλίνης. Είστε συνδεδεμένος, μπορούμε να σας ακούσουμε, παρακαλώ. Καλό απόγευμα από το πολύπαθο και φιλόξενο νησί της Λέσβου. Θέλω να πω ότι η Λέσβος έχει σηκώσει όλο αυτό το μεταναστευτικό, το σφυγικό ζήτημα που ταλανίζει το νησί και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μια πενταετία. Οι Λέσβοι πολίτες άνοιξαν μια μεγάλη αγκαλιά, στάθηκαν αλληλέγγυοι απέναντι στους μετανάστες, όμως οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για το νησί της Λέσβου ήταν πολύ μεγάλες έχει φτάσει πια, έχει εξαντληθεί η ενδοχή των κατοίκων του νησιού μας, έχει διαλυθεί η κοινωνική συνοχή και βέβαια οι οικονομικές, όπω είπα, περιπτώσεις όχι μόνο των πολιτών αλλά και του ίδιου του Δήμου είναι πολύ μεγάλες. Είμαστε εδώ για να διατυπανίσουμε και να διαμηνήσουμε σε όλους ότι νιώσαμε πολλές φορές και συνεχίζουμε να νιώθουμε μόνοι. Δεν είναι δυνατόν η Λέσβος η οποία έχει σηκώσει τις πλάτες στο σύνολο του μεταναστευτικού ζητήματος και βεβαίως έχει ζήσει πολλά επεισόδια που τελευταία αυτό το κάψιμο το κιτ της Μόργερς με αποτέλεσμα οι μετανάστες να έχουν αυτή τη στιγμή εγκατασταθεί σε μία δομή η οποία είναι τελείως κατάλληλη μέσα στον αστικό ιστό της πόλης με πολλές επιπτώσεις οι οποίες θα έχουν και συνέχεια. Εν μέσω πανδημίας δεν είναι δυνατόν να συνοστίζονται 7.000 άτομα και πλέον μέσα σε μια υποτυπώδη δομή. Είναι επιβεβλημένο να γίνει άμεσα μια γενναία αποσυμφώρηση και να καταλάβουν και οι φίλοι μας Ευρωπαίοι ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι όχι μόνο προς τους μετανάστες αλλά και προς τους κατοίκους της Λέσβου. Ας καταλάβουν όλοι ότι η ίση κατανομή και η αλληλεγγύη μεταξύ μεταναστών και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών αυτή τη στιγμή είναι επιβλημένη. Ας καταλάβουμε όλοι ότι τα σύνορα της Λέσβου και το νησιό μας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα πρέπει να φυλάξουμε όλοι για να διαφυλάξουμε και τα κεκτημένα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ας καταλάβουμε όλοι ότι οι ΜΚΟ, οι, οποίοι, οι οποίες έχουν ελεγχθεί ως ένα μεγάλο βαθμό τελευταία από την ελληνική κυβέρνηση, όλες δεν επετέλεσαν το σκοπό τους αλλά πολλές από αυτές είχαν ιδιωτελείς σκοπούς. Έχουν καυθεί ενδιστάσεις στον κόσμο, έχουν καυθεί ενδιστάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε χάσει τη συνοχή μας και βέβαια οι επιπτώσεις στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ας καταλάβουμε λοιπόν, επιμένω, ότι θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε τα νησιά μας, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου όπως τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο οι οποίες υπέστησαν πολλά δεινά πανδημία, μεταναστευτικό και τελευταία ο σεισμός. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Είμαστε αλληλέγγυοι απέναντι σε όλους όσοι στέκονται με ορθολογιστική σκέψη απέναντι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει όλους μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όπως έχουμε κάνει στη συνέχεια ε, βοηθώντας στο να γίνει μία δομή, ένα κέντρο ταυτοποίησης, ολιγομελές, εκτός κατοικημένης περιοχής και έξω από αστικό της πόλης και το οποίο θα πληρεί όλες τις συνθήκες Ασφάλεια και υγιεινή τόσο για τους ίδιου τους μετανάστες, όσο και για τους συμπολίτες Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτή τη βάση να κινηθούμε για να κλείσουν όλες οι υπόλοιπε δομέ, οι οποίες είναι πλέον 7 μέσα στο Δήμο μυτιλήνης και το λέω αυτό γιατί ο Δήμος μυτιλήνης φιλοξενεί το σύνολο των μεταναστών στο νησί της Λέδρα. Θα πρέπει λοιπόν να εγκαινοθούν κάποια σπίτια στα οποία φιλοξενούν ε, μαζικά μετανάστες υπό άγνωση συνθήκης υγιεινής και ασφάλειας και να μαζευτούν όλοι σε μία δομή η οποία θα είναι ελεγχόμενη και θα πληρεί τους κανόνες ασφάλειας και για άλλους λόγους, και για άλλους λόγους εκτός από αυτούς και για λόγους εθνικούς. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθηθούμε να ενισχυθούμε οικονομικά γιατί έχουμε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά και οι αντοχές μας πλέον έχουν εξαντληθεί. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Μητυλίνης αλλά και το οικονομικό πακέτο του Δήμου πηγαίνει για να εξυπηρετήσει το μεταναστευτικό ζήτημα. Με αποτέλεσμα πολλές δομές να έχουν μείνει πίσω στο Δήμο Μητυλίνης αλλά και άλλες να έχουν διαλυθεί still... Κύριε Κιτσέλη, αν θέλετε ολοκληρώστε, γιατί έχουμε να ακούσουμε ακόμα και τον Δήμαρχο της ε, Λαμπεδούζας και να ε, συνεχίσουμε. αλλά ζητάμε επίσης την επίσκεψη του ταυτοποίησης ασύλο έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται άσυλο να μείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπόλοιποι να πάνε πίσω στα σπίτια τους από εκεί οι οποίοι μας ήρθαν. Ε, αυτά ήθελα να καταθέσω, βάζω στην αγωνία όλων των κατοίκων του Αιγαίου και βεβαίως ας καταλάβουν και οι φίλοι μας Ευρωπαίοι ότι το ζήτημα είναι όλων μας και όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, τα περιμένει στη φωτιά και στο δικό σα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Thank you, Mr. Vitalis. Now let's hear from Salvatore Martello. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μαρτέλο. Προσπαθείτε να περιοριστείτε σε τέσσερα λεπτά για να έχουμε χρόνο και για τους υπόλοιπους ε, ομιλητές και μετά να ακούσουμε και τους προσκεκλημένους μας, την κυρία Γιώχανσον, τον ε, κύριο Σιχόφερ και τον κύριο Χρήστο. Κύριε Μαρτέλο, δήμαρχε της Λαμπεντούζα, ευχαριστώ. Η Λαμπεντούζα, το νησί μου, είναι 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα με περίπου 1500 κατοίκους στο κέντρο της Μεσογείου και είναι γνωστή σε όλη τη Μεσόγειο όχι μόνο γιατί είναι το νησί που βρίσκεται στα πλέον νότια άκρα της Τύρου μας αλλά γιατί φτάνουν διαρκώς ε, σκάφη με μετανάστες στο νησί. Εδώ και 30 χρόνια έχουμε τέτοιου είδου ε, αφήξεις. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κατεπίγουσα ανάγκη τεράστιων διαστάσεων και ε, αυτό που έχει δημιουργηθεί στο νησί, όποιος δεν το έχει δει δεν μπορεί να το φανταστεί. Στην Λαμπεντούζα οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί και από την πανδημία του COVID-19. Η Λαμπεντούζα είχε εγκατεληθεί στην τύχη της ακόμη και όταν ήταν απαραίτητο να υπάρξει απτή βοήθεια από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο σύμφωνο. Τα λόγια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπογράμμισαν την πρόθεση να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Όμως ταυτόχρονα το σύμφωνο, ε, ε, επιμένει στις επιστροφές και ε, αφήνει να παραμείνουν οι μετανάστες που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγες. Εδώ το θέμα δεν είναι αν θα διασώσουμε κάποια ανθρώπινη ζωή, αλλά ποιε θα είναι οι αρχέ ε, στου οποίου θα βασιστούμε. Χρειάζονται μηχανισμοί πραγματική διάθεση που να επιβαρύνουν το ίδιο όλα τα κρατημέλη. Ε, είδαμε μια πολλωστή δραματική περίπτωση ναυαγίου στη Μεσόγειο πρόσφατα. Και Είδαμε να χάνει τη ζωή του ένα παιδί 6 μηνών έξι μηνών και στην πορεία του από την Αφρική προς τα τελικά κατέληξε σε ένα τάφο στην κοταφείο της Λαπεντούζα. Αυτά είναι τα θλιβερά που ζούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα. Όταν μιλάμε για τις επιστροφές ε, υπάρχουν ενδιασμοί. Σήμερα στην Λαμπεντούζα ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει υγειονομικός έλεγχος για τον COVID και οι υπόλοιπε διαδικασίες ελέγχου ε, έχουν Υπάρχουν σοβαρέ καθυστερήσει από τι μεταφορέ από τα σκάφη καραντίνα και την εξέταση στα διάφορα hotspot του νησιού. Ε, δυσκολεύεται η λειτουργία των hotspot και βεβαίως χρειάζεται απαραίτητη ταξινόμηση των ε, μεταναστών που είναι δύσκολο αν ε, χαρακτηριστούν είτε πρόσφυγες είτε οικονομικοί μετανάστες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ε, θα είναι θέμα λοιπόν τη ταχύτητα τη διαδικασία, ο χαρακτηρισμό του κάθε ανθρώπου και σκεφτείτε για τις περιοχές των ε, συνόρων. Ε, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργούνται ανοιχτοί καταβλισμοί μεταναστών, πόσο ε, επισφαλείς είναι οι συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν. Όμως υπάρχει και το θέμα του τουρισμού. κυρία ε, Φοντερ επενήχθηκε ότι θα πρέπει να το θεωρήσουμε τελειωμένο αυτό το θέμα. εδώ πρέπει να ε, προληφθούν μέτρα στήριξη των νησιών που βρίσκονται στα σύνορα. Για τα ανατολικά και τα νότια της Ευρώπης πρέπει να ληφθεί κάποια μέρημνα, διότι ε, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε πώς θα, θα θωρακίσουμε και τη Λαμπεντούζα και άλλα 19 ακροπύργια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εάν δεν υπάρξουν απλώς ε, οι σωστές επιστροφές και περιορίσουμε την παρουσία ε, προσφύγων, θα πρέπει να δούμε ότι ένας αριθμός, μικρός αριθμός των μεταναστών, σίγουρα έχουν δικαίωμα να παραμείνουν εδώ, αλλά θα είναι δύσκολο επίσης να εφαρμοστεί ένα μηχανισμό των επιστροφών. Πρέπει να γίνεται όλα αυτά σε κάθε περίπτωση με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υπάρξουν νόμιμοι για όσους θέλουν μια καλύτερη ζωή και τίποτε παραπάνω. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι στους κανόνες που θα προβλέψουμε για την μετανάστευση. Θα υπάρχει πάντοτε και ε, θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά με ανθρωπιά. Γιατί δεν εμποδίσουμε τις ροές των μεταναστών, θα πρέπει κυρίως να τις διαχειριστούμε καλύτερα και να τις διοργανώσουμε. Στην ε, Λαμπεντούζα με την ε, αφοσίωση και τη δουλειά των τοπικών κυβερνήσεων και των πολιτών έχουμε ε, βασιστεί στους στόχους ε, του ΟΗΕ για την νόμιμη και ελεγχόμενη, ρυθμιζόμενη μετανάστευση. Εδώ χρειάζονται φάνταστες ε, καινοτόμες λύσεις, διότι δεν αρκεί να καταργήσουμε κάθε αρχή διάσωσης ανθρώπινων ζώων αλλά να βρούμε μια λύση ρεαλιστική. Και μια τελευταία πτυχή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχω χρόνο, ήθελα απλώς να πω ότι για το σχετικό μανιφέστο χρειαζόμαστε ασφαλείς οδούς μετανάστευσης διότι στην Λαμπεντούζα προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, όποιον μπορούμε αλλά να παραμείνει και το νησί ένα νησί που δεχόμαστε ε, όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και τουρίστες. Ευχαριστούμε και προσπαθήστε να μας υποστηρίξετε σε αυτόν τον δρόμο. Ευχαριστούμε Δήμαρχε Μαρτέλο. Χαίρομαι που άκουσα νέα από τη Λέσβο και από τη Λαμπεντούζα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή αυτή μας συζήτηση. Ε, πραγματικά το καυτότερο ζήτημα, η πιο επικίνδυνη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ότι έχουμε 600 αφήξεις τη μέρα ε, πάνω από 2.000 τα Σαββατοκύριακα. Ε, έχουμε μια σειρά από παράγοντες που επιβαρύνουν το φαινόμενο λόγω της πανδημίας στην Αφρική και βλέπουμε και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξύνουν την κατάσταση. Αναστολή των προγραμμάτων μετακατάστασης, ε, μηχανισμοί αλληλεγγύης στομωμένοι Και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται κατεπηγόντω. Να περάσουμε τώρα στου υπόλοιπου αγορητέ μα και μετά η προσκεκλημένο μα. Η κυρία ε, Καρίνη Φάρα. Mr. Lopez Aguilar, Mrs. Karimi is not connected. Η κυρία Καρίνη δεν είναι συνδεδεμένη, κυρία Αγγιλάρ. Ντάνιελ Μιλεύσκη τότε. Not connected. Δεν είναι συνδεδεμένος. Πιέτρο Μάρτολο. Συνάδελφε, είστε συνδεδεμένος. Με ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα είναι πυλώνες επί των οποίων πρέπει να βασιστεί η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη για μένα είναι μία και μόνη. Ε, θα πρέπει η κατανομή των ευθυνών να ε, μην έρχεται πάντοτε σε αντιδιαστολή με τον ανθρώπινο πόνο αυτών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να, ε, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Βλέπουμε πώ χαρούν τη ζωή του προσπαθούν να φτάσουν ω εδώ. Ε, Δεκάδε χιλιάδε ετούντε άσυλο ζουν σε συνθήκε απάνθρωπε. Αυτού του είδου την αλληλεγγύη θέλουμε. Αυτό ήθελα να διαβάσω στο σύμφωνο ότι αλλάζει. Και κυρία Επίτροπε, να σα πω, γιατί δεν είχατε την τόλμη να προτείνετε ένα σύστημα μόνιμη μετα... με σε υποχρεωτικό και διαρκέ. Γιατί δεν προτείνατε ένα μηχανισμό συντονισμού για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα. Χρειάζεται ε, να ε, διαφωνήσετε ενδεχομένω με τα κράτη-μέλη και να επιβάλλετε μέτρα, αλλά όχι για την αναχέτηση, για την καλή διοργάνωση που αντλούν από τι θετικέ πτυχέ τη μετανάστευση. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να το πετύχουμε χάρη και στην επιρροή του Κοινοβουλίου και σε διαπραγματεύσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε τη σπαραχτική κραυγή μια μάνα που χάνει το παιδί τη ε, και να βλέπουμε τι ζουν στους καταβλισμούς ε, οι άνθρωποι στη Λιβύη για να φτάσουν στην Ευρώπη. Και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Τι τύχη θέλουμε να έχουν οι άνθρωποι αυτοί που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παραμένουν και πρέπει να επιστραφούν. Ε, αυτοί που θα ζουν ε, σε παράνομες συνθήκες ε, στα κράτη-μέλη είναι καλύτερο να ζήσουν σε συνθήκες κράτησης σε τρίτες χώρες. Όχι κυρία Επίτροπε, δεν είναι αυτή η αλληλεγγύη για την οποία έχει αγωνιστεί η Ευρώπη. Δεν ζούμε εδώ ε, και σας μιλάω εδώ από τη Λαμπεντούζα. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Επόμενος. Τόμας Μπάλασεκ, αν είναι συνδεδεμένος. Όχι, δεν είναι συνδεδεμένος. Not connected. Not connected. And Thierry Mariani. Not connected. Connected. Then we will try Did leave you Brailo. Not connected, but we have now... Um... Δεν έχει συνδεθεί κανεί από όσου έχετε φωνάξει, αλλά έχουμε τον κύριο Μπράνκο, λέει η συντονίστρια. Ποιος? Γκριν Μπράνκο. Α, μάλιστα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Hello. Ναι, με ακούτε. Μπορείτε παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε την κάμερα. see me now? but we can hear you if you speak in English. Δεν θα μεταφραστεί ο κύριος Μπράνκο εάν δεν έχει κάμερα. Βάλτε την κάμερα παρακαλούμε. Στον. Για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και να μεταφραστείτε. Αλλιώς δεν θα μεταφραστείτε. It's okay now. Oh, hello. Τώρα είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα. Εμείς θεωρούμε ότι από κοινού πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει όμως η Ευρώπη να προασπίσει τα εξωτερικά της σύνορα. Δεν χρειάζεται μαζική μετανάστευση Ευρώπη. Χρειάζεται μια πραγματική πολιτική για τις οικογένειες, για τους πολίτες των χωρών της. Η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα. Και βρίσκεται σε σημαντική γεωστρατηγική θέση. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε σε όλα τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη πως η παράτυπη αυτή μαζική μετανάστευση θα επιδεινώσει την κατάσταση και τα προβλήματα. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Ρεαλιστικά πρέπει να ενεργήσουμε και όλοι από κοινού. Παραβάνω χωρίς ε, μεγαλώστομες δηλώσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Προβλήματα που δεν τα έχουμε δημιουργήσει εμείς, δεν τα έχουμε προκαλέσει. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να δώσουμε ένα τέλος και αυτό πρέπει να κάνουμε. μόνο όσοι χρειάζονται πραγματικά άσυλο πρέπει να βοηθηθούν. Επίση, οι χώρε προέλευση πρέπει να βοηθηθούν, οι χώρε προέλευση των ανθρώπων αυτών, για να μπορούν εκεί να είναι ασφαλεί, να μπορούν να εργαστούν, να έχουν ε, τα προστοζήν. και όχι να έρθουν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την Ευρώπη που είναι ήδη επιβαρημένη, αντιμετωπίζει από πλευράς ασφάλειας ε, μια τραγική κατάσταση Συν αυτή την κατάσταση ασφάλειας έχουμε τώρα και την πανδημία. Πανδημία και μετανάστευση. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε σαν αυτό να μην είναι πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Η Ευρώπη ε, θέλει ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Να επανέλθει η Ευρώπη στις βασικές της αξίες, που είναι η συνεργασία, η ασφάλεια και ο αλληλοσεβασμός. Όμως το σλόγγαν μας θα πρέπει να είναι πρώτα η Ευρώπη, πρώτα οι Ευρωπαίοι, οι παραδόσεις των Ευρωπαίων, ο πολιτισμός ο ευρωπαϊκός. Μία Ευρώπη υπάρχει μόνο. Thank you. Thank you so much. If there no other speakers... Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, θα πρότεινα να δώσουμε εκ νέου το λόγο στους διακεκριμένους προσκεκλημένους του πάνελ για να μας δώσουν τις αντράς. Καταρχάς η κυρία Γιώχανσον. Κυρία Επίτροπε, ακούσατε τα σχόλια όσων μπόρεσαν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση γιατί όπως διαπιστώνετε έχουμε πολλά προβλήματα σύνδεσης. Τα βίωσε και ο κύριος Ζέχοφερ, ε, εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας ε, της Εκπεριτροπής Προεδρίας της Ένωσης. Κυρία Γιώχανσον, κάποια σχόλια αν έχετε την καλοσύνη. Commissioner, please press speak. Η κυρία Επίτροπος να πατήσει το κουμπί Speak. Παρακαλούμε. Κύριε Επίτροπε, είστε εκεί. Όχι, χάσαμε την επαφή μας. Να την ξαναβρούμε μήπως. Να προσπαθήσουμε ή τον κύριο Ζέιχόφερ. Είστε εκεί, είστε έτοιμος. Sie haben Äh, να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν ειδικά τους δύο δημάρχους και το πώς τον ε, ε των γιατρών χωρίς σύνορα. Να πω ακόμη μια φορά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κρίνεται στα εξωτερικά σύνορα ποιος ε, πρέπει να τύχει προστασίας και ε, μπορεί μετά να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος δεν ε, δικαιούται προστασία πρέπει να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Και εδώ και εμείς και η Κομισιόν ε, συνάπτουμε συμφωνίες ε, με τις χώρες προέλευσης έτσι ώστε να μπορούμε και να βοηθήσουμε εκεί αυτούς τους ανθρώπους. Αναφέρθηκαν και οι διαπραγματεύσεις για την ε, δήλωση με την ε, Τουρκία. Νομίζω ε, μπορεί να γίνει και με άλλες χώρες. Μιλάμε για τα δύο τρίτα των μεταναστών, τα οποία ούτε με το εθνικό ούτε με το διεθνές δίκαιο δικαιούνται προστασία. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται προστασία θα πρέπει να κατανεμηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ελληνική και Βεβαίως. Ε, αντιλαμβάνομαι και άλλες μορφές της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της, πρό... πρότασης της Κομισιόν με την οποία συμφωνούμε ως Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι μια ανθρωπιστική απάντηση η Ευρώπη με τις θεμελιώδεις αξίες της προσφέρει στους ανθρώπους οι οποίοι διώκονται και φοβούνται για τη ζωή τους προστασία και αυτό το στηρίζουν και οι λαοί της Ευρώπης κατά πλειοψηφία. Με το σημερινό σύστημα δεν γίνεται αυτό. Έτσι θα έχουν λυθεί τα δύο τρίτα των προβληματικών περιπτώσεων. Δεύτερον, χρειαζόμαστε νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης για αυτούς οι οποίοι ε, αναζητούν εργασία στην Ευρώπη για οικονομικούς λόγους και οι περισσότερες χώρες ε, και η δική μου χώρα χρειάζονται ε, εργαζόμενους. Ε, ποια είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή. Αν δούμε το τι γίνεται στις χώρες αύξησης ε, στην Λαμπεντούζα και στη Λέσβο. Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει η εγγύηση ότι δεν θα παραμένουν εκεί οι πρόσφυγες αλλά θα κατανέμονται με τρόπο αλληλέγγυο στην Ευρώπη. Αυτή είναι θεμελιώδης αρχή και ε, βλέπω ότι μένει εκτός των συζητήσεων. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς που χρειάζονται προστασία και να μην έχουμε έναν εξέλιγκτο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη γιατί έτσι θα χάσουμε την στήριξη των λογικών ε, ανθρώπων. Ήμουν ε, και πρωθυπουργός της Βαβαρίας ε, ή τώρα είμαι υπουργό ε, της Γερμανίας. Ε, αυτά που σας λέω προκύπτουν από την εμπειρία μου. Θα ήθελα να πω τον Δήμαρχο Λέσβου πως έχουμε πάρει σχεδόν 2.000 ασυνόδευτούς ανηλίκους και οικογένειες στη Γερμανία. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει ήδη έρθει και προς τον Δήμαρχο της Λαμπεδούζας θα ήθελα να πω πως η Γερμανία πάντα συμμετείχε στην υποδοχή ε, ατόμων που ε, από την Μεσόγειο στην Ιταλία. Δυστυχώς στην κατανομή αυτή συμμετέχουν έξι, το πολύ 7 ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την εισδοχή των ατόμων αυτών. Για να αλλάξει αυτό ακριβώς εκεί πέρα στοχεύει η πρόταση της ε, Κομισιόν. Ε, την οποία στηρίζουμε. Δηλαδή να προστατεύσουμε όσους δικαιούνται προστασία, οι υπόλοιποι να επιστρέψουν, Αμέ μην τους αφήσουμε στην τύχη τους να συμφωνήσουμε με τις ε, χώρες προέλευσης ε, και τελικά να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή λύση για όσους διασώζονται θάλασσα δεν υπάρχει θέμα αλλά ε, μέχρι στιγμή πολύ λίγε χώρε ε, το δέχονται, όλοι οι υπόλοιποι δεν το δέχονται. Γι' αυτό χρειάζεται επιγόντω μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση. Και να πω ακόμη μια φορά, εάν δεν το καταφέρουμε ε, το προσεχέ μέλλον, τότε οι ακραίοι αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικρατήσουν και πέρασα ολόκληρη την πολιτική μου ζωή έτσι ώστε οι ακραίοι, ειδικά από τα δεξιά, ε, να μην ε, ε, κάνουν κουμάντο στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια στιγμή κρίσιμη όπου δεν έχει νόημα μόνο να λέμε τη λέξη αλληλεγγύη. Είναι εύκολο αυτό. Πρέπει να γίνουν οι συμφωνίες, να ληφθούν οι αποφάσεις για να γίνει κιόλας. Και συχνά στην Ευρώπη είχαμε μεγάλες αποφάσεις. Την διεύρυνση προς Ανατολάς σε πολλά ζητήματα. Πάντα είχαμε την δύναμη να τα λύσουμε αυτά. Και βασίζομαι ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Ja, sehr geehrter. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ μπορούμε να επιστρέψουμε τους συναδέλφους εφόσον θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Οπότε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία το λόγο στην κυρία Λουίζα Άμσπεργκερ από την ε, Γερμανική Μοσπονδιακή Βουλή. Ευχαριστώ για την δυνατότητα ε, να τοποθετηθώ και εκ μέρους των Πρασίνων της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις, επικριτικές ίσως, από κοινοβουλευτικής σκοπιάς. Μας ανησυχεί πολύ το θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε για την κατάσταση όπως έχει ε, διαμορφωθεί στην Ευρώπη και για το κατά πόσον η πρόταση που έχει γίνει μέσω του συμφώνου είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι τελώς άγνωστο εάν θα εγκριθήκαν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και τι θα γίνει ε, με την ε, Μεσόγειο και τις περιοχές της και αυτό είναι ένα βασικό σημείο επίκρισης. Μετά είναι το θέμα της ευθύνης καθημερινά βλέπουμε ε, να υπάρχουν ε, τέτοια θέματα στην καθημερινή επικαιρότητα και να απασχολούν την κοινή γνώμη. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τι έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Όλα αυτά μας ε, φέρνουν σε μια θέση που μας αναγκάζουν να περασπιστούμε τις ευρωπαϊκές ε, αρχές μεν, αλλά πρέπει από κοινού ε, να τις προασπιστούμε. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει και επιπλέον ήδη τώρα πρέπει να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μιλήσουμε ε, ειλικρινώς και δήμος ε, ε, μεταξύ μας. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή και πραγματικά απευθύνω μια απελπισμένη έκκληση προς τον κύριο Ζιχόφερ, προς όποιον μπορεί να κάνει κάτι και με ακούει, ήδη τώρα να φροντίσουμε να μην ποινικοποιηθεί περαιτέρω η διάσωση στη θάλασσα και να ε, διαφυλάξουμε αυτή την ευρωπαϊκή αξία. Ανθρώπινε ζωέ πρέπει να διασώζονται ε, στην θάλασσα. Αυτό είναι το πρώτο. Και μετά το δεύτερο είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασία των Συνόρων. Ε, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν και εκείνοι τι δικέ του ευθύνε. Είναι μια κινητήριο δύναμη. Αυτή έχει γίνει τώρα. Αλλά βλέπουμε πώς, μπορούν, πώς προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν και να το χειραγωγήσουν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη μεταναστευτική Πολίτη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε μόνο από κοινού να τη διαμορφώσουμε και να την εφαρμόσουμε πραγματικά ε, συνδυάζοντας τις ε, απαραίτητε ε, ανάγκες. Για αυτό το θαυμάσιο ελληνικό νησί και τα υπόλοιπα πέραν της Λέσβου πρέπει να εργαστούμε μαζί και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να πετύχουμε την προστασία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Μαριανή. Τιερή Μαριανή, είστε συνδεδεμένος. Δεν βλέπω καμιά απάντηση. Ο κύριος Λίβιου, Χάιλιου ε, είναι συνδεδεμένος. Πατήστε το speak παρακαλούμε. Να του δώσουμε το λόγο. Is having some Έχει προβλήματα σύνδεσης. Ίσως προχωρήστε και να επανέλθουμε. Ο κύριος Έρικ Μάρκετ. Έρικ Μακάρ. Δυστυχώς ακούμε ελάχιστα τον ομιλητή Εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε την κατάσταση λίγο στα χέρια μας, να μην περιμένουμε τις έτοιμες προτάσεις Επιτροπής και Συμβουλίου. Είδαμε τι έχει γίνει ε, στο νησί της Λέσβου. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε μια κατάσταση να διονύζεται. Πιστεύω ότι επίσης δεν μπορούμε να επικρίνουμε τον κόσμο ότι απλουστεύει τα πράγματα ως προς τη μετανάστευση. Κάποιοι πάντοτε θα κατηγορούν ε, γιατί δεν είναι όλοι άξιοι διεθνούς προστασίας. Πρέπει όμως να δούμε εμείς τις κατάλληλες διαδικασίες και στα σύνορα. διότι βλέπουμε ότι επί τόπου είναι πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν ε, ad hoc. Κάποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν έγγραφα, άλλοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν και να αποφασιστεί αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή όχι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες και αυτό είναι σημαντικό να περάσει ως πρόταση. Ε, εδώ στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο συζήτηση πέραν αυτής της διάσκεψης ε, και το τι θα υποθεί στα κράτη-μέλη στην Επιτροπή. Θα πρέπει να επιδιώξουμε να προχωρήσει η όλη αυτή η συζήτηση και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Αυτή είναι η δική μας ε, ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να μην συνεχίσουμε να αναβάλουμε την εξέφραση λύσεων. Ευχαριστούμε και να ακούσουμε και τον τελευταίο αγόρτη, τον κύριο Μπέρναρ Μπέκερ, εάν είναι συνδεδεμένος. Από τι κάτω χώρες, Μπέρναρ Μπέκερ. Auch nicht? Ούτε εσεί. Δεν είναι σταθερή η σύνδεση. Τότε να δώσω το λόγο στην κυρία Γιώχανσον, γιατί δεν έχουμε πλέον χρόνο, και θα παρακαλέσω την κυρία Γιώχανσον εάν μπορεί ε, να απαντήσει στις ερωτήσεις όποιος προλαβαίνει και να κάνει και μια καταληκτική παρέμβαση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό που μίλησαν οι δήμαρχοι ε, από τη Λέσβο και τη Λαμπεντούζα μακάρι να μπορούσαν να πάρουν και άλλοι βουλευτές το λόγο, αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση. Για να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάνουν προσπάθειες να σώσουν ε, ανθρώπινες ζωές ε, στη θάλασσα και δεν πρέπει να ποινικοποιούνται σε καμία περίπτωση. Και αυτό προτείνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε δημοσιοποιήσει πριν από δύο μήνες. Τώρα, ε, ο ΕΑΣΟ που ελπίζουμε ότι θα γίνει ένας οργανισμός ασύλου αλλά και η Frontex είναι οι δύο αυτοί φορείς που βοηθούν από, το γάμα από τη γάμα δέλτα home και τη δική μου γενική διεύθυνση. Επίσης είναι άνθρωποι εκεί που βοηθούν τον κόσμο στα ελληνικά νησιά, στη Λαμπεντούζα και στα Κανάρια νησιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι ετέθησαν πολύ σημαντικά ζητήματα για την ανάγκη εξέβρεση ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύη και ευθύνη, αλλά αυτό που επίση κάποια από εσά αναφέρετε, μια ισορροπία μεταξύ επιστροφών και μετακαταστάσεων. Και αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Δεν θα πρέπει δηλαδή να ε, ρηψοκινδυνεύουν οι άνθρωποι μέσα από πάρα πολύ ε, αντίξωες συνθήκες ε, ένα ταξίδι προς την Ευρώπη. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποφύγουμε το να, τους να αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να καταφύγουν ε, σε αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν πρώτον να ε, αποφύγουν τη διακίνηση ε, κυνηγώντα τους διακινητές ε, και να βοηθήσουμε και στις χώρες προέλευσης. Όσοι δεν είναι τώρα επιλέξιμοι να παραμείνουν, όσοι δεν είναι πρόσφυγες, πρέπει να επιστρέψουν, πρέπει να επιστραφούν. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον που δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό άχθος τα μικρά νησιά που είναι και το, ο τόπο πρώτη άφηξη των ανθρώπων αυτό. Πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Εξού και προτείναμε οι συνορικές διαδικασίες για τις οποίες είμαστε υπέρ, να γίνονται στα σύνορα και μόνο αν είναι ε, ανάγκη ε, να γίνονται στην ενδοχώρα, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια ανάγκη, γιατί ε, πράγματι αναγνωρίζουμε την πολύ δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλά ελληνικά νησιά. Τώρα που δεν υπάρχουν πολλές αφήξεις, και βλέπουμε ε, σίγουρα ότι φτάνουν ίσως ε, περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες θα πρέπει τις παράτυπες αφήξει ε, να τις περιορίσουμε και αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Λέλη. Σας ευχαριστώ κυρία Γιωχάνσον και τώρα για να ολοκληρώσουμε θα κάνω και εγώ την τελευταία δήλωσή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επιτροπό, τον Υπουργό τον κύριο Ζεχόφερ, τους δύο δημάρχους, ε, τον κύριο Χρήστο και όλους τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό το πάνελ. Είδαμε ότι ήταν λίγο δύσκολο τεχνικά, αλλά υπήρξε καλή βούληση και ευχαριστώ και τους συμμετέχοντες εύχομαι στον κύριο Ζεχόφερ και στην κυρία Ιωχάνσεν καλή δύναμη για τις τελευταίες εβδομάδες γερμανικής προεδρίας και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την κοινή πολιτική ασύλου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει. Ευχαριστώ πάρα, πολλούς, ε, πάρα πολύ όσους βοήθησαν στην συζήτηση και βεβαίω έχουμε μετά και τον επόμενο γύρο. Well, I think we're coming close to the... Νομίζω πλησιάζουμε στο τέλος. Ήταν αρκετά μεγάλη πρόκληση γιατί έχουμε διάφορες ε, δυσκολίες, ε, λάθη στην επικοινωνία, πρόκληση και για τους ομιλητές όπως και να έχει ε, έγινε μια συζήτηση και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες υπό τις συνθήκες της πανδημίας που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, ως δήλωση θα έλεγα ότι η μετανάστευση είναι γεγονός. Δεν μπορεί να είναι πρόκληση για μια τεράστια δύναμη και στην οικονομία και σε όρους νομικούς ε, και ηθικούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το αντιμετωπίσει. Η μετανάστευση είναι γεγονό δεν μπορεί να είναι βάρος ε, ε, δυσβάσταχτο, όχι για τα 27 κράτη-μέλη της ε, Ένωσή τη. ούτε για κάθε ένα από τα ω μέλος της. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιο κράτος μέλος μόνο του, ούτε κάποιο κράτος να μην κοιτάει τα εξωτερικά σύνορα όταν έχουμε μια μαζική είσοδο όπως είδαμε και στην ε, Λαμπεντούζα που μας είπε ο Δήμαρχος ο κ. Μαρτέλο ή στη Λέσβο όπως μας είπε και εκεί ο Δήμαρχος ο κ. Σκητέλης ε, ή στα Κανάρια αυτή τη στιγμή όπου η αίσθηση είναι ότι τα νησιά μένουν μόνα τους ε, και ακριβώ ε, και πάλι αμφισβητείται η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι λοιπόν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται όταν ε, υπάρχει αυτό το αίσθημα ε, στους απλούς ανθρώπους, στις εθνικές τοπικές αρχές που ζητάνε ελεγγύη και κοινή ευθύνη. Μεγάλες προσδοκίες λοιπόν υπάρχουν Σύμφωνα αυτό. Και βεβαίως μιλάμε και για αυτούς τους ανθρώπους ε, στις ε, ΜΚΟ που προσπαθούν να διασώσουν, να μειώσουν τους θανάτους ε, και στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, στα Κανάρια, όπου υπάρχουν πολλοί θάνατοι σε καθημερινή βάση. Πολλοί περνάνε, αλλά πολλοί δεν τα καταφέρνουν. Πολλοί πεθαίνουν στην προσπάθεια να φτάσουν ε, στα εξωτερικά σύνορα. Είτε είναι τα ε, νησιά στο Αιγαίο, είτε τα Ιταλικά νησιά, είτε η Καναρίνηση. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές ε, τις δυσκολίες, θα τις ξεπεράσουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τις συζητήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ.